Ωραία. Περνάμε στο δημόσιο τμήμα τη ακρόασή μα. Α εγκρίνουμε καταρχήν την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντίρρηση για τη σημερινή ημερήσια διάταξη, α την εγκρίνουμε παρακαλώ. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Όπως ξέρετε δεν μεσολάβησαν ολομέλειες ε, στο Στρασβούργο από την τελευταία μας συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου, εκ τούτου δεν έχουμε κατεπήγοντα ψηφίσματα. Να σας υπενθυμίσω ότι την επόμενη 3η 6 Σεπτεμβρίου θα γίνει η ετήσια η μας συνάντηση με τους ε, επικεφαλής αντιπροσωπιών, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Ευρωπαίους πρέσβεις. Οπότε παρακαλώ Δώστε το παρόν για την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους εκπροσώπους μας που μας βοηθούν πολύ και είναι απαραίτητοι για το έργο μας στο εξωτερικό και μας βοηθούν και στις αποστολές και τις αντιπροσωπείες που πραγματοποιούμε ανά τον κόσμο. Θα ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση με ένα τμήμα που θα γίνει υπό την Προεδρία του Πρόεδρου Σούλτσα και παρουσία της ΥΠΑ της εκπροσώπου Μογκερίνη από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα στις 6 Σεπτεμβρίου. Επόμενο θέμα. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 30 Ιουνίου 2016. Υπάρχουν ερωτήσεις, ε, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, όχι, οπότε εγκρίνεται. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, για να ε, μην υπερβούμε το χρόνο μας, γιατί όπως ξέρετε η διερμηνία έχουμε μέχρι τις 12.30, θα περάσουμε στο σημείο 7, τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και σε άλλες γειτονικές χώρες, της Ανατολικής, εταιρι... Ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και άλλες γειτονικές χώρες. Θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Παντσέρη ε, προς την έκθεση της Επιτροπής ΦΑΜ με το ίδιο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Παντσέρη για το έργο του το σχέδιο γνωμοδότησης ήδη έχει μεταφραστεί και το έχετε λάβει. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η διορία για την υποβολή των τροπολογιών λύγει την επόμενη Πέμπτη, την επόμενη Δευτέρα, συγγνώμη, 5 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι. Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου. Κύριε Παντσέρη, παρακαλώ, έχετε 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να διευκρινίσω καταρχήν ε, το εξής, ότι στην επικεφαλίδα ε, της ε, αυτής ε, γίνεται λόγος για τα δικαιώματα των γυναικών στην ανατολική, με την ανατολική εταιρική σχέση και όχι με άλλες χώρες. Εγώ θέλω να συμβάλλω στην έκθεση που έχει συσταθεί σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και αναφέρομαι κυρίως ε, στη ε, ζωή των γυναικών ε, στις ανατολικές χώρες, στην ανατολική εταιρική σχέση, σε χώρες που βρίσκονται στην ανατολική εταιρική σχέση. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι γυναίκες αυτές κατά τη διάρκεια της μετασυγκρουσιακής περίοδου δεν μπόρεσαν να διαδραματίσουν ρόλο σε επίπεδο κυρίως ε, συνδικαλιστικό. Βεβαίως ε, θα έπρεπε να υπάρχει μια οριζόντια προσέγγιση έτσι ώστε να ενταχθούν και αυτές σε όλες τις ε, τομέκες πολιτικές, σε όλες τις πολιτικές της, των γειτονικών χωρών, των ανατολικών γειτονικών χωρών. Ένα άλλο θέμα είναι η εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες στις ανατολικές γειτονικές χώρες πολλές φορές εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να συνεχίζουν σε ανώτερη ε, εκπαίδευση. Και αυτό καταδεικνύει λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να ξεπεραστούν τα νομικά κολλήματα έτσι ώστε να επικρατήσει τελικά, ε, να επικρατήσουν ίσες ε, συνθήκες αμοιβών η έκθεση επίσης κάνει έκκληση στις ανατολικές μας χώρες να επικυρώσουν την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Ε, απευθύνεται κυρίως σε χώρες που δεν το έχουν κάνει. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σεξουαλική βία, στην παράνομη διακίνηση ανθρώπινων όντων. Αυτά πλήττουν κυρίως ε, τις ε, ευαίσθητες περιοχές, τις γυναίκες και κυρίως εκείνες ε, που βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη. Και τέλος, εγώ αναφέρομαι στην πλατφόρμα του Πεκίνου που γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην σεξουαλική και άλλη ζωή των ε, ε, γυναικών. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, έχουν ήδη καθοριστεί οι προθεσμίες για να κατατεθούν τροπολογίες. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η δική μας άποψη την οποία και θα καταθέσουμε στην Επιτροπή Γυναικών. Σας ευχαριστούμε κύριε Παντζέρη. Θέλει κανείς το λόγο από τους και οδησίτες. Η κυρία Σόιντροβα και μετά ο κύριος Αυστρεβίτσιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, της ε, υποεπιτροπής ε, που θα δοθεί για την έκθεση της Επιτροπής Γυναικών για τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τις άλλες γειτονικές χώρες. Η Επιτροπή Γυναικών δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το αντικείμενο, το περιεχόμενο της έκθεσής της, οπότε θα σχολιάσω μόνο τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή και εκτιμώ ιδιαίτερως ε, τις βασικές ιδέες και την πρόταση της πολιτικής ανάμειξης ε, των γυναικών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και την οικονομική τους χειραφέτηση. Επίσης, ε, Συμμερίζομαι την άποψή σας για την ανάγκη να αποστεύσουμε τις γυναίκες από βία, εμπορία και εκμετάλλευση. Επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γειτονικές μας χώρες να εξασφαλίσουν καλύτερη μόρφωση των γυναικών και να δώσουν έμφαση στην παιδεία των κοριτσιών και καθώς και στην καλύτερη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες και θα κάνω κάποια σχόλια. Καταρχήν, η γενική απέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής σταθερότητας στις χώρες αυτές είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση. Επίσης, έχω κάποιες πιο λεπτομεριακές ε, τροπολογίες ε, που θα τις υποβάλω στον εισηγητή. Αφορούν την παιδεία, την επιχειρηματικότητα, την απασχολησιμότητα, την υγειονομική φροντίδα και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Δεν συμφωνώ με το άρθρο 11 που είναι υπερβολικά ε, μακροσκελές και αφορά την πρόσβαση ε, των γυναικών ε, στις υπηρεσίες που αφορούν την ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Θα κάνω σχετικές τροπολογίες. Αυτά εν συντομή ήταν τα σχόλιά μου και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία ώστε η γνωμοδότησή μας να συμπεριληφθεί στην έκθεση της Επιτροπής Γυναικών και μάλιστα πλήρης. Ευχαριστώ για την έκθεση και προσβλέπω στη συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Σόιντροβα. Ο κύριος Αυστρεβίτσιος. Σας ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Παντσέρη για τη γνωμοδότησή του και ε, είναι πολύ χαρά, μεγάλη χαρά για μένα το να είμαι σκιώδη σε αυτή την έκθεση, όχι να τον επισκιάζω, αλλά να είμαι σκιώδης συνεργάτης του. Όσον αφορά λοιπόν στην ενσωμάτωση της διάστασης ε, του φύλου ε, και την μη διακριτική μεταχείριση είναι καθοριστική σημασίας ε, στη διαδικασία μεταρρύθμισης να συμπεριληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να ελέγχουμε ε, τις, ε, τα επιτεύγματα κατά τα επόμενα έτη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις που αφορούν σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ε, οι τροπολογίες των φιλελευθέρων θα κατατεθούν εν ευθέτω χρόνο. Ξεκινάω λοιπόν και θέλω να σας πω ότι οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αλλά όπως και άλλες χώρες οι γυναίκες που ζουν σε αυτές τις χώρες πρέπει να συμμετέχουν με τους ίδιους όρους ε, σε όλες τις ε, διαδικασίες. Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να επιδεικνύουν ηγετική πολιτική πυγμή ε, σε όλες τις εκφάνσεις της ε, ζωής και αυτό είναι ένα ε, ηχηρό και ουσιαστικό ε, σημείο κίνησης για τη γνωμοδότησή μας. Επιπλέον, η κοινωνική και η οικονομική εξουσιοδότηση, η απόκτηση εξουσίας αυτούς του δύο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι οι γυναίκες να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και εάν χρειάζεται να είναι και καλύτερα ενημερωμένες. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι η βοήθεια που προσφέρεται, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράμματα συνεργασίας, η βοήθεια αφορά ακριβώς αυτό που προανέφερα. Και τέλος πιστεύω ότι και αυτή η γνωμοδότηση θα συμπεριλαμβάνει τροτές ομάδες όπως είναι οι γυναίκες με αναπηρία. Αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ξανασχοληθούμε. Γιατί πολλές χώρες, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Παντσέρη, ασχολούνται με γυναίκες με τα συγκρουσιακά καθεστώτα. Κυρία Πρόεδρε, με όλα αυτά κατά νου, νομίζω ότι τελικά θα έχουμε μια καλή γνωμοδότηση από την ε, Επιτροπή μας και η δική μας ομάδα των φιλελευθέρων θα συμμετέχει ουσιαστικά. Πρόεδρος, εάν ε, λοιπόν... Ε, Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτινς που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε με τον εισηγητή. Καλωσορίζουμε και την έκθεση αυτή, καθώς και τις συστάσεις. Η ενδοοικογενειακή βία, η διακριτική μεταχείριση λόγω φίλου, ε, είναι θέματα που εξακολουθούν να ε, ε, μας απασχολούν σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Επίσης, η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών παραμένει χαμηλή. Ε, είναι στα πατριαρχικές μες, στερεότυπα κλισέ, φαλοκρατικά τα οποία περιορίζουν την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, στην, ε, ακόμη και στην κοινωνική ζωή, στην αγορά εργασίας. Για την συγκεκριμένη περίπτωση της Ουκρανίας, επειδή υπάρχει η σύγκρουση, βλέπουμε ότι πλήττονται κυρίως όπως προς τις μαζικές εκτοπίσεις, κυρίως ε, οι γυναίκες και τα παιδιά. Ε, στις 20 ε, Ιουλίου είχαμε τελευταία έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι υπάρχει ο διάλογος με τις έξι χώρες ανατολικής γειτονίας και Αναφερθήκαμε με αυτό το ζήτημα του ε, ε, συνδρόμου μετά από σοβαρό τραύμα, ε, σοβαρή τραυματική εμπειρία όλων όσων επιστρέφουν από εμπόλεμες ζώνες για την υποχρεωτική διάγνωση και αποτελεσματικές θεραπευτικές αγωγές για όλα τα μέλη της οικογένειας. Αυτό είναι συγκεκριμένα για την Ουκρανία, αλλά όπως σας είπα στα πλαίσια του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που γίνεται και με τις έξι χώρες της πολιτικής γειτονίας, Ανατολική γειτονία. Ε, φέτος είχαμε και με τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία επίση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του διαλόγου έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο για την ισότητα των δύο φίλων και την ενδοοικογενειακή βία. Παρακολουθούμε λοιπόν εκ του συνεγγύς το ζήτημα και ενθαρρύνουμε τις χώρες εταίρους να θεσπίσουν νομοθεσία για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και κυρίως για να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της νομοθεσίας προτείνει επέκταση των δικών της συστημάτων, ε, στρατηγικές και σχέδια δράσης που ήδη υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, αναφέρθηκε ε, νωρίτερα, πέρα από την νομοθεσία, είναι νομικά όργανα που διαθέτουμε και ε, συνεχίζουμε μια τη δέσμευσή μας για την αρρωγή προς τα, τις χώρες της πολιτικής ανατολικής γειτονίας. Είναι μέχρι τη μερίμνα της υπηρεσίας μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαρτά, ο κύριος Παντσέρη. Θέλετε να κάνετε και τα τελικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Θα είμαι ε, σύντομος. Ευχαριστώ για τις, ε, τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα δύο-τρεις ε, διαστάσεις του Δήματος μόνο να σχολιάσω. Η ο Σοντρόβα το τόνισε και συμφωνώ και εγώ. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, να επισημάνουμε πως υπάρχει σχέση και με τη σταθερότητα στη χώρα. Ε, και ε, είναι σίγουρα ε, θετική οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε και για τη σταθερότητα της περιοχής. Στην, στο σημείο 11 είναι ξεκάθαρο από τη συζήτηση ότι υπάρχουν διαστάσεις απόψεων η χρησιμοποίηση της πλατφόρμας του Πεκίνου, παραδείγματος χάρη, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και επί τη βάση των τροπολογιών θα συσκεφθούμε και πάλι και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική συμβαστική λύση. Ευχαριστώ επίσης κυρία Οστρεβίτσιους. Μπορώ να υποστηρίξω αυτά που είπατε για την συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω ρόλος του ε, και νομίζω ότι μπορούμε να εξεργαστούν περισσότερο αυτά τα στοιχεία που σχετίζονται με το θέμα. Ε, η επόμενη ημερομηνία είναι η 26 Σεπτεμβρίου, τότε θα μπορέσουμε να συναντηθούμε και για τις ε, τροπολογίες μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να αποφασίσουμε από κοινού. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχιστούν οι επαφές και οι συζητήσεις μας. Α, ακριβώς κύριε Παντσέρη, σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας. Ε, Ήσασταν πολύ συγκεκριμένοι στις ερωτήσεις σας, κάνατε εύστοχα ερωτήματα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ευχαριστούμε και πάλι την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την παρουσία τους. Ευχαριστώ και τα μέλη που ήταν εδώ. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ.